E Καλημέρα συνάδελφοι. Ο κύριος Μάουρος ζητάει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρεμβαίνω βάσει του 173 άρθρου του κανονισμού. Απόψε τη νύχτα το ανώτατο δικαστήριο της Βραζιλίας αρνήθηκε την, την πέλαση του ε, δολοφόνου Τσέζαρε Μπατίστη. Δύο ψηφίσματα του Κοινοβουλίου μας είχαν ζητήσει να υπάρξει μια απόφαση ή απέλεση προς την Ευρώπη. Θέλω να εκφράσω πέρα από τη λύπη μου ε, την επιθυμία η Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εκφράσει τη λύπη ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη δυσαρέσκεια του έναντι των Βραζιλιανών αρχών και να εκφράσουμε Επίσης την αλληλεγγύη μας προς τις οικογένειες των δολοφονημένων που εδώ και 30 χρόνια περιμένουν δικαιοσύνη. Ευχαριστώ κύριε Μάουρο. για αυτήν τη σωστή σας παρατήρηση. Παρακαλώ συνάδελφοι, κύριε Μποργέτσιο να τελειώνουμε. Η λύπη εκφράζεται από όλο το κοινοβούλιο όπως και η πίκρα για τις ε, λιμένες αποφάσεις. Εγώ δεν μπορώ παρά να επαναλάβω όλα όσα το Κοινοβούλιο εξέφρασε για δύο φορές με τα ψηφίσματά του. Με αυτή λοιπόν τη θλίψη και με αυτήν τη σαφήνεια θα διαβιβάσουμε προς τις αρχές της Βραζιλίας την λύπη μας. Ροντζούλη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Με δύο δευτερόλεπτα. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Βάισμπεργκερ που είναι εδώ με το μωρό της ε, και που είναι νεογέννητο, όπως επίσης και σε όλες τις νεομαμάδες αυτού του κοινοβουλίου που με δυσκολία μπορούν να είναι καλές μαμάδες και καλές βουλευτίνες. Θα ήθελα να το εκφράσω αυτό ως σύμβολο ελπίδας. Προσοχή, είναι σημαντικό και πραγματικά με καίει. Λοιπόν, να δω αν θα σοβαρευτείτε λίγο. Σας παρακαλώ. Άκουσα δυστυχώς αυτές τις μέρες φράσεις αυτού του στυλ. Το κοινοβούλιο δεν είναι παιχνιδότοπος, δεν είναι νηπιαγωγείο. Έξω τα παιδιά και έξω οι μανάδες τους. Και επίσης η παρουσία παιδιών ε, προσβάλλει την εικόνα του Κοινοβουλίου. Επειδή εμείς προσπαθούμε εδώ να συνδυάσουμε η οικογένεια και δουλειά, ε, είναι λυπηρό και σχρόν ακούγονται τέτοιες φράσεις στο Κοινοβούλιο. Διότι εμείς αυτό προσπαθούμε να συνδυάσουμε, την οικογένεια με τη δουλειά μας. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν στην ημερήσια διάταξη πριν ψηφίσουμε. Θέλω να κάνω εδώ μερικές δηλώσεις. Ανακοινώσεις καλύτερα. Πρώτη, γραπτή δήλωση 007-2011 που παρουσίωσαν οι κύριοι Παπαστάμκος, Μπεναχμίας, Μίτσελ, Σούστα και Σύρκα